Επίτροπε, έληξε η συζήτηση. Διακόπτεται και η συνεδρίαση. Θα συνεχιστεί αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Σας εύχομαι καλή νύχτα.